ιστορία, έχει πολιτισμό. Και δεν μιλάμε μόνο για ένα απλό χρηματοδοτικό εργαλείο. Το InvestEU πρέπει να είναι φαλτήριο προς μια Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ε, ακολουθεί αυτές τις αλλαγές και θα οδηγήσει σε αυτή την αλλαγή ε, παραδείγματος. Θα πρέπει επίσης να είμαστε προοδευτικοί είναι μια Ευρώπη που θέλουμε να δημιουργήσουμε, που θα είναι κοντά στους πολίτες, δίνοντας συγκεκριμένες ελπίδες και φιλοδοξία. Πάκετ. Πρόεδρε, Ευχαριστώ, θα μπορέσουμε να επενδύσουμε στην καινοτομία. Περίπου 40 δισεκατομμύρια με τη μορφή δεν πρόκειται για επιχορηγήσεις, πολλές επενδύσεις θα μπορέσουν να υλοποιηθούν σε πολλούς τομείς. Οι ευρωπαϊκές εταιρείε θα τύχουν υποστήριξη και θα μπορέσουν να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα. Δεν θα εξαρτώνται από εξωευρωπαίους δωρητές. Θα γίνει μια σύμπηξη λοιπόν των εφισταμένων χρηματοδοτικών επενδυτικών μηχανισμών. Αυτό είναι εξαιρετικό. Τα πάντα πλουστεύονται οι εθνικές προθερικές τράπεζες αποκτούν σημαίνοντα ρόλο. Οι φλεμμαδικές τράπεζες θα έχουν σημαίνοντα ρόλο και στη δική μου χώρα. Πιστεύω ότι το αποτέλεσμα λοιπόν είναι έκτακτο, έξοχο. Η αλλαγή αυτή θα φέρει αποτελέσματα. Πρόκειται για την τελευταία μας ολομέλεια βεβαίω. και πιστεύω ότι τελειώνουμε πραγματικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρους της ομάδας Άλντε, κυρία Βίρινγκ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Αγαπητοί συνάδελφοι, Είχαμε καταρχάς το ΕΦΣΙ και τώρα το InvestEU, το οποίο θα δραματίσει ένα σημαντικό ρόλο και στην επόμενη θητεία. Και δείχνει μια πολύ σημαντική κατεύθυνση. Ένα από τα διδάγματα που αντλήσαμε από την κρίση του 2008 είναι ότι η σταθερή οικονομία συνιστά ε, μια οικονομία των επενδύσεων. 650 σε, σε παραπάνω επενδύσεις λόγω του προγράμματος. Και αυτό είναι μια υπόσχεση για το μέλλον.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 για την επίτευξη ικανοποιητική συμφωνία όσον αφορά τα βασικά στοιχεία του προγράμματος InvestEU. Όπω είπε και η Επίτροπο, παρέχουμε ένα κίνητρο, ενθάρρυνση στις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν με το επόμενο κοινοβούλιο. Έχουμε ξαναμιλήσει για το πρόγραμμα αυτό, γιατί όντω πρόκειται για πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία όμως θα έχει η μελλοντική εφαρμογή στα κρατημέλη. Θα πετύχει όταν γίνει πιο ορατό, όταν κατορθώσει να χρηματοδοτήσει έργα τα οποία δεν μπορούν να χρηματοδοτηθούν από εμπορικές τράπεζες ή από το Ταμείο Συνοχής. Εμείς όμως πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην κοινοτομία, στις νοφείς επιχειρήσεις, Πρέπει να τις βοηθήσουμε να μεγαλώσουν σε μέγεθος. Πρέπει να βοηθήσουμε όλους τους επιχειρηματίες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και οι οποίοι αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία. Ας επενδύσουμε λοιπόν σε έργα τα οποία έχουν μια δυναμική, τα οποία μας δεν εκτιμά η αγορά. Χρειάζεται επίσης προσοχή στην γεωγραφική κατανομή των πόρων. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων αφορούσε κυρίως τις πιο χώρες. Ήρθε η ώρα όμως να βοηθήσουμε και τις άλλες. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρο, ευχαριστώ. Κύριε Περέση, παρακαλώ. Ένα μισή λεπτό. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, η έγκριση του κειμένου εντάσσεται στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προκρίθηκε με το σχέδιο Juncker και, την, και πίεση των σοσιαλιστών. Είναι μερική η νίκη μας εν ώψη της περίοδου 21-27 ε, αλλά χαιρόμαστε έστω και γι' αυτό. Όσον αφορά την διακυβέρνηση, σίγουρα έχουμε πετύχει μια καλύτερη ισορροπία, διότι υπάρχει μια διευθύνουσα επιτροπή, μια επιτροπή διακυβέρνησης, όπου συμμετέχει και η Κομισιόν και άλλοι θεσμικοί εταίροι, εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το νέο αυτό πρόγραμμα θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις κλειδί με οικολογικό επίσης σκοπό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αγκαλιάσει το θέμα των αηφορικών υποδομών, των επενδύσεων στην κοινωνία και στις δεξιότητες καθώς και στον τομέα του πολιτισμού. Προσοχή όμως, το θέμα της καλύτερης στοχοθεσίας. Πρέπει να σταθούμε στο ύψος των δεσμευσεών μας πρέπει το 40% των επενδύσεών μα να πάει προ το πρασίνισμα τη οικονομία. Και να θυμηθούμε και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για άλλη μια φορά τη δίνει προεξέχοντα ρόλο. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για καλή απόφαση όσον αφορά ε, τα δικαιώματα που θα έχει στην κατεύθυνση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. παρακαλώ. E αφορά κυρίως τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Παρά κάποιες ενστάσεις που έχω και στις οποίες θα αναφερθώ στο τέλος. Το θέμα είναι λοιπόν να εγγυηθούμε τον στόχο της αντιμετώπισης της μεταφορίας του κλίματος. Το θέμα είναι καλύτερες συμβουλευτικές υπηρεσίες, καλύτερη γεωγραφική κατανομή. Λήψη υπόψη της ανάγκης προστασίας του κλίματος Τώρα, ως προς τις συναστάσεις μου, βλέπω ότι εντάσσεται το πρόγραμμα μας και η άμυνα, καθώς και άλλα έργα τα οποία δεν έχουν σχέση με την προστασία του κλίματος. Βλέπω αεροδρόμια, βλέπω επενδύσεις στην ενέργεια μέσω των ρηκτών καυσίμων. Θέλουμε να κάνουμε κάτι για το μέλλον του πλανήτη ή όχι. Όταν έρθει ο Μάιος λοιπόν και η ώρα των εκλογών, σκεφτείτε τι ανάγκε του πλανήτη. Πρόεδρος. Ε, ο κύριος Πασπισίλη έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι συναδελφοί μου ε, με κάλυψαν ήδη λέγοντα πολλά σημαντικά πράγματα όσον αφορά το πρόγραμμα Invest in You, το οποίο προφανώ υποστηρίζω. Θεωρώ ότι το παιδιτικό αυτό πρόγραμμα είναι πολύ σημαντικό. Η εμπειρία που είχαμε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων έχει δείξει ότι οι πρωτοβουλίες αυτές είναι απόλυτα λογικές, σκόπιμες και ότι είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να επικεντρωνόμαστε μέσω επενδύσεων σε τομεί οι οποίοι δεν χρηματοδοτούνται αρκετά. Χαίρομαι πάρα πολύ που το πρόγραμμα Invest in Youth επικεντρωθεί στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Χαίρομαι πολύ που θα προωθήσει τους στόχους αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών, θα προωθήσει τους περιβαλλοντικούς στόχους και την πολιτική έρευνας και καινοτομίας. Πιστεύω ότι στο μέλλον το πρόγραμμα InvestEU θα προωθήσει εν γέννη την ευρωπαϊκή οικονομία, ακριβώς επειδή έχει ένα, μπορεί να έχει πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι παρέχει εγγύησεις για ιδιωτικά δάνεια. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω λοιπόν το διάδοχο πλέον του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Θεωρώ ότι έχουμε αντλήσει πολύ θετικά διδάγματα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και χαίρομαι πάρα πολύ που θα έχουμε και την κατάλληλη χρηματοδότηση από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021 με 2027. Ευελπιστώ λοιπόν ότι το επόμενο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην επόμενη θητεία θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα αυτό ώστε να αρχίσει να υλοποιείται από το 2020 και μετά. Κύριος Φερνάντες, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Πριν πέντε χρόνια οι σοσιαλιστές όταν κατεβήκαμε στις ευρωεκλογές απαιτούσαμε το τέλος ε, της λιτότητας ε, των πολιτικών προσαρμογής ε, και ζητούσαμε να δοθεί μεγαλύτερη τόνωση και όθηση στις επενδύσεις για να ξεπεράσουμε την κρίση. Φυσικά και ευχαριστούμε και την Κομισιόν και όλες τις πολιτικές ομάδες που προώθησαν το σχέδιο Juncker γιατί αυτό ήταν σημαντικό για να αντιμετωπιστεί τα τελευταία χρόνια η κρίση. Και είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε το βήμα που γίνεται τώρα για τη δημιουργία ενός μόνιμου εργαλείου. Το νέο αυτό Invest Europe, Invest EU, που θέλει να συνεχίσει να τονώνει τι επενδύσει ε, και να τη στηρίζει μόνιμα στην Ένωση είναι κάτι πολύ απαραίτητο αυτή τη στιγμή που βιώνουμε μια μεγάλη περίοδο στασιμότητας και τελμάτωσης. Ε, το σχέδιο Γιούνκερ, ε, όμως ε, εξακολουθεί να χρειάζεται αντικυκλική πολιτική, όπως αυτή που μπορεί να προσφέρουν αυτά τα προγράμματα. Ευχαριστώ κύριος Μπούντα. Ένα μισή λεπτό. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητέ. Το πρόγραμμα InvestEU είναι μία από τις ε, πιο κεντρικές πλέον πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωση, που είναι σε θέση να κινητοποιήσει εγγυημένε ιδιωτικές επενδύσεις. Και κατά αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα πολύ πιο φιλικό προβλέψιμο κλίμα για τους επενδυτές. Και βέβαια κατά αυτόν τον τρόπο μέσω των επενδύσεων αυτών συμβάλλουμε στην ευημερία των πολιτών μέσω καλύτερης οικονομικής και κοινωνικής σύγκλησης, μέσω της έρευνας, της καινοτομία, της ψηφιοποίησης και μέσω της υπεύθυνη χρήση των πόρων. Επί του παρόντος, οι επενδύσεις βλέπουμε ότι επικεντρώνονται σε ορισμένα μόνο κράτη-μέλη. Μέσω του προγράμματος αυτό InvestEU και μέσω των επιλέξιμων προγραμμάτων θα είμαστε σε θέση να πετύχουμε την κατάλληλη γεωγραφική ισορροπία προκειμένου να μην αυξάνονται περισσότερο ανισότητε μεταξύ των περιφερειών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, α μην στο ξεχνάμε ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει δραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συνήθω αντιμετωπίζουν πολύπλοκε διαδικασίε όταν, όταν προσπαθούν να εξασφαλίσουν επενδύσει. Έρχεται λοιπόν τώρα το πρόγραμμα Invest in You για να απλουστεύσει τι διαδικασίε αυτέ και να μειώσει τη γραφειοκρατία σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, θα πρέπει να καταφέρουμε να προσελκύσουμε επενδύσει, ιδίω σε κάποια μικρά τοπικά προγράμματα, ακριβώ εκεί που μπορεί να επιτευχθεί μόχλευση και εκεί πέρα που μπορούν να συμμετέχουν πολλά κλάστερ ε, επενδυτών. Οι δημόσιε όμω αρχές θα πρέπει και πάλι να διασφαλίσουν ότι θα υπάρχει απαραίτητη δανειοδότηση και το απαραίτητο θετικό ε, κλίμα προκειμένου να προσελκυθούν περισσότερε επενδύσει. Κύριε Ρούμπιχ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Κάρας ε, της, ε, του Intergroup για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ο οποίος στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρόκειται για πάρα πολύ σημαντική στρατηγική απόφαση, γιατί θέλουμε να πετύχουμε την ευημερία τους πολίτες και μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Εδώ και 25 χρόνια ξέρω πολύ καλά τι ε, έχουν πετύχει τα ΔΕΛΤΑΠΗ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 500 δις ε, διατέθηκαν και από το 2007 στο 2013 που προωθήσαμε το πρόγραμμα για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα με 2 δις. Και βέβαια έχουμε και το Micro ΜΜΕ, 3 δις και το εύση με 500 περίπου ε, δις μαζί με τη μόχλευση. Έτσι λοιπόν σε ευρωπαϊκό επίπεδο δείχνουμε ότι λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας την ανάγκη να στηρίξουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το 25% τώρα ε, προβλέπεται για επενδύσεις στον τομέα του κλίματος. Ε, και βλέπουμε ότι έχει κάνει έτσι μία στροφή προοδευτική η Ευρωπαϊκή Όνωση για να ε, είμαστε πρωταγωνιστές ε, και θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο Μπιενκόφσκα γιατί γνωρίζω ότι δεν είναι εύκολο ε, να στηρίξει κανείς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δείξαμε όμως ότι αυτό είναι εφικτό. Ευχαριστώ και καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ. Διαδικασία προσέλκυσης προσοχής ε, του Προέδρου Κάτς Διάη. Μία, ε, ένας μάλλον ιστισόλογο, κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το πρόγραμμα InvestEU πράγματι θα μπορούσε να αποδώσει και θα μπορούσε να συμβάλλει πραγματικά στην ανάπτυξη, στη δημιουργία θέσεων εργασίας, να στηρίξει την κατάρτιση, να στηρίξει τις δεξιότητες αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αποφύγει τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν με το σχέδιο juncker διότι η εμπειρία από το ευρωπαϊκό ταμείο στρατηγικών επενδύσεων ιδίως για την ελλάδα απέδειξε ότι τον πακτολό των χρημάτων τον πήραν οι ευρωπαϊκές πολυεθνικές οι οποίες στην πράξη χρηματοδοτήθηκαν για να αρπάξουν τα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας. κλασική περίπτωση η fraport η οποία υποτίθεται ότι θα έκανε επενδύσεις στο πλαίσιο μιας δίθεν αποκρατικοποίησης που επέβαλε η τρόικα και έχουμε μια κρατική γερμανική εταιρεία η οποία παίρνει δάνειο 280 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλα τόσα από Ελληνική Τράπεζα και αρπάζει τα περιφερειακά αεροδρόμια. Τέτοιου είδους επενδύσεις δεν νομίζω ότι συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. Απλά χρηματοδοτούνται οι δίθεν ιδιωτικοποιήσεις άρα λοιπόν το πρόγραμμα πρέπει να πάει σε μια κατεύθυνση στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με αυξημένη προστιθέμενη τοπική αξία. ευχαριστώ. Ε, σας ευχαριστούμε πολύ και τώρα δίνω το λόγο στην ε, κυρία Μπιενκόφσκα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί βουλευτέ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συζήτηση αυτή, καθώς και για τα θετικά σας ε, σχόλια για το πρόγραμμα και το βασικό συμπέρασμα το οποίο συνάγω από αυτή τη συζήτηση είναι ότι υπάρχει συντριπτική υποστήριξη ε, υπέρ του προγράμματο InvestEU. Πάντως σημειώνω βέβαια και τι πολύ ψηλέ προσδοκίε σα και τις συστάσεις σας ε, για την εφαρμογή αυτού του προγράμματος και θέλω να σας πω ότι θα τις μεταφέρω και θα τις λάβουμε υπόψη αυτές τις συστάσεις ε, κατά την προπαρασκευή του προγράμματος. Ξανά να ευχαριστήσω τους συνεισηγητές αλλά και όλους όσοι λάβατε το λόγο. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε πολύ και για να ολοκληρώσουμε θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή κύριο Φερνάντες. Οι δημόσιε επενδύσει ε, είναι πάρα πολύ σημαντικέ. Οι ιδιωτικέ επενδύσει εξίσου σημαντικέ. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την ιδιωτική πρωτοβουλία, να τονώσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ένωσης, ε, την επιχειρηματικότητα, τις νεοφύης επιχειρήσεις, να ενισχύσουμε την ε, παραγωγικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό σημαίνει ότι θα αμείβονται καλύτερα, με καλύτερους μισθούς, οι εργαζόμενοι και στο δημόσιο αλλά και στον ιδιωτικό τομέα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ό,τι αφορά τώρα τις δημόσιες επενδύσεις, είναι πάρα πολύ σημαντικό οι κυβερνήσεις ε, να κάνουν τη δική τους δουλειά. Δυστυχώ στη χώρα με την Πορτογαλία. Με το τρέχον επενδυτικό πρόγραμμα, η κυβέρνηση και ιδίω ο Πέδρο Μάρκε, ε, ο αρμόδιο υπουργό, δεν έδωσαν ούτε ένα ευρώ ε, για επενδύσεις. Το έργο, το σχέδιο Juncker και το InvestEU θα πρέπει να αξιοποιηθούν για δημόσιες επενδύσεις μεταξύ άλλων, όχι μόνο για ιδιωτικέ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι να βάλουν το λιθαράκι τους. Ε, στο κοινοβούλιο αυτό εγκρίναμε αυτό το πρόγραμμα. Μιλάμε για 700 ε, δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία κινητοποιούνται. Πάρα πολύ καλή γεωγραφική κατανομή. Έτσι ε, ενισχύουμε και αυτή την πλατφόρμα, αυτό το συμβουλευτικό κόμβο του InvestEU. Πρέπει να υπάρχουν όμως σε εθνικό επίπεδο τέτοιοι κόμβοι που θα βοηθούν τους επενδυτές. Θα μπορούσαν να είναι και περιφερειακές βέβαια οι πλατφόρμες αυτές ε, με στόχο να βοηθήσουμε να διαρθρωθούν τέτοιου είδους επενδυτικές πλατφόρμες και να ε, κατατίθενται καλές υποψηφιότητες για την αξιοποίηση του InvestEU. Εγώ είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε περισσότερη ε, σε επενδύσεις, μεγαλύτερη οικονομική ανάπτυξη, απασχόληση, πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Θα πετύχει δηλαδή ε, τους στόχους του αυτό το πρόγραμμα του InvestEU. Ευχαριστώ πολύ. Και στο πέρα τη θέλω να ευχαριστήσω όλους για την συνεργασία. Οι ψηφοφορίες θα λάβουν χώρα αύριο. Θα είναι και η τελευταία μας συνεδρίαση. Ξεκινούμε στις 8 και μισή έως τις 2. Η μέση διάταξη είναι ήδη δημοσιευμένη στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βλέπω τον κύριο Ρούμπιχ όμω που θέλει τον λόγο. Ναι κύριε Πρόεδρε, εξ ονόματος ε, των ε, βουλευτών που είναι παρόντες θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί προεδρεύατε υποδεγματικά πάντοτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Και ελπίζω και υπό άλλες συνθήκες να ξανασυναντηθούμε κατηδίαν ίσως και να έχουμε και άλλες τέτοιες συζητήσεις στην ωραία σας τη χώρα. Ευχαριστώ και πάλι ο Πρόεδρος. Και κλείνει η συνεδρίαση εδώ σε αυτό το σημείο.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 διακοπή σα συνεδρίαση. Τα χθεσινά πρακτικά και τα κείμενα που έχουν εγκριθεί είναι στη διάθεσή σας. Παρατηρήσει αν δεν υπάρχουν, εγκρίνονται τα πρακτικά. Και περνούμε στο πρώτο σημείο της απογευματινής μας ημερήσιας διάταξης. Έκθεση Μετσόλα, Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Η κυρία Μετσόλα, η συγγήτρια, έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ανατέθηκε σε μένα η έκθεση αυτή και κανείς δεν φανταζόταν ε, ότι θα καταφέρναμε έξι μήνες μετά την υποβολή της πρότασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντάξουμε την έκθεση αυτή. Χρειάστηκε λοιπόν να καταβάλουμε πολλέ προσπάθειες, χρειάστηκε να αναλύσουμε όλε τι τεχνικέ πτυχέ και λεπτομέρειε τη πρόταση αυτή, χάρη όμω την ιδιαίτερη επικοδομητική συνεργασία που είχαμε του συναδέλφου εδώ στο Κοινοβούλιο, με τα κράτη-μέλη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταφέραμε να συμφωνήσουμε επί ενό νέου συστήματο για το οποίο μπορούμε να είμαστε όλοι περήφανοι. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων είχαμε κατά νου ότι θα πρέπει να είμαστε δίκαιη απέναντι σε αυτούς οι οποίοι χρειάζονται προστασία, αυστηρή με όσου είναι παράτυποι μετανάστες και ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί και απαιτητικοί με όσους εκμεταλλεύονται του πιο ευάλωτους ανθρώπους. Θέλουμε να επιβεβαιώσουμε λοιπόν τώρα τη νέα αυτή νομοθεσία και σε αντίθεση με ό,τι θα περίμενε κανείς αρχικά καταφέραμε να επερκεράσουμε όλα τα προβλήματα και καταλήξαμε τελικά σε μια νέα πρόταση για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Θεσπίσουμε συγκεκριμένο αριθμό συνοριοφυλάκων, προκειμένου να μπορούμε πραγματικά να διασφαλίζουμε την ασφάλεια των εξωτερικών μας συνόρων, προκειμένου να μπορούμε να καταπολεμούμε την διεθνή εγκληματικότητα και προκειμένου να μπορούμε να διασφαλίζουμε τα δικαιώματα όσων χρειάζονται προστασία και προκειμένου να μπορούμε βέβαια να διαχειριζόμαστε και τη μετανάστευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολύ σημαντικό τα κράτη-μέλη να έρθουν στο ύψο των ευθυνών του. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο το νέο αυτό σύστημα το οποίο προτείνουμε αυτή τη στιγμή θα είναι αποτελεσματικό. Βέβαια, η νομοθεσία αυτή δεν είναι η μοναδική λύση που χρειαζόμαστε στον τομέα τη μετανάστευση, είναι καθοριστική όμω σημασία προκειμένου να καταφέρουμε να συνδυάσουμε την νομοθεσία αυτή με τι υπόλοιπε νομοθεσίε. Αν αντιμετωπίσουμε ανάλογη κρίση με αυτή που είχαμε το 2015, τότε τα κράτη-μέλη τα οποία βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα, όπω η Μάλτα ή πολλέ άλλε χώρε, θα μπορούν πλέον να έχουν επιπλέον προσωπικό και θα μπορούν πλέον να έχουν την απαραίτητη συνδρομή την οποία χρειάζονται για να αντιμετωπίσουν αυτέ τι καταστάσει κρίση. Η νομοθεσία λοιπόν αυτή που έτυχε διαπραγμάτευση στους τελευταίους μήνες δεν αφορά μόνο τα 10.000 αυτά επιπλέον άτομα. Σημαίνει επίσης ότι μπορούμε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα του συστήματος επιστροφής για όσους είναι παράτυποι μετανάστες. Μα δίδονται με τη νέα αυτή νομοθεσία περισσότερε δυνατότητε να συνδράμουμε τα κράτη-μέλη, ιδίω όσον αφορά τον εντοπισμό των παράτυπων μεταναστών και μπορούμε επίσης μέσω της νέας αυτής πρότασης κανονισμού να μπορούμε να δώσουμε, να χορηγήσουμε πιο εύκολα συνδρομή προ του νόμου μετανάστε και να του δώσουμε και τα απαραίτητα εξωτικά έγγραφα. Έχουμε νέε αρμοδιότητε πλέον για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή. Μπορεί πλέον ο οργανισμό αυτό να προασπίζει και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων θα πρέπει να προστατεύονται. Απότερο στόχο μα είναι να έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο προστασία, το οποίο να συνάδει με τι βασικέ ευρωπαϊκέ αξίε, οι οποίε για μα είναι πάρα πολύ σημαντικέ, ιδίω για ένα τόσο ευαίσθητο θέμα. Και αυτό διότι βέβαια γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό τη θα πρέπει να προασπίζει τα θεμελιώδη δικαιώματα. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ο Επίτροπο κ. Αβραμόπουλο έχει τώρα το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, στη γλώσσα σας ε, σας ευχαρίστησα. Πώς ήταν η προφορά μου. Θέλει λίγο ακόμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, Δεν σας κρύβω ότι τα σύνορα και η ακτοφυλακή είναι ένα βασικό βήμα για μια συνολική πολιτική μετανάστευση. Δημιουργήσαμε και εγκαταστήσαμε και ενισχύσαμε σε χρόνο ρεκόρ τον οργανισμό αυτών με κοινέ προσπάθειες. Γνωρίζοντας πολύ καλά τη συνθετότητα των νομοθετικών διαδικασιών συμφωνούμε όλοι ότι πρόκειται περί κατορθώματος. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την εισηγήτρια κυρία Μέτσολα και όλους τους σκιώδεις και τη Ρουμανική Προεδρία που ε, κατέληξαν σε ισορροπημένη συμβιβαστική λύση επί της πρότασης. Η συμφωνία υπογραμμίζει πάλι ότι, και πάλι όταν συνεργαζόμεθα έχουμε καλά αποτελέσματα και δείχνουμε στους πολίτες ότι η Ένωση είναι πρόθυμη και ικανή για δράση. Όταν η, κρίση κορυφώθηκε στην Ευρώπη το καλοκαίρι του 2015, η Ευρώπη ε, κατελήφθη εξαπίνης και δεν ήταν έτοιμη. Αντιμετωπεί με εισρωή παράτυπων ε, εισόδων από Ανατολάς και Νότο, από τη Μεσόγειο, ε, καταλάβαμε ότι έπρεπε να αναλάβουμε αποφασιστική δράση. Δεν υπήρχε ε, ο ενιαίος οργανισμός για τα σύνορα, ούτε υπήρχε, υπήρχαν επιχειρησιακές ικανότητες επιτόπου. Το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου δεν ήταν κατάλληλο για αυτή τη δουλειά. Τα συστήματά μας πληροφόρησης δεν μιλούν, συνομιλούν μεταξύ τους και οι προσπάθειές μας ε, για να εντάξουμε τρίτες χώρες ήταν κατακαιρματισμένες. Αναγκαστήκαμε να λάβουμε άμεσα μέτρα και μακροπρόθεσμα μέτρα και να εργαστούμε παράλληλα σε όλα αυτά τα μέτωπα. Τώρα, τέσσερα χρόνια αργότερα, Όποιος ε, προσπαθήσει να περάσει παράτυπα τα εξωτερικά μας σύνορα εντοπίζεται, ε, λαμβάνονται δακτυλικά αποτυπώματα και εξετάζεται σε βάθος. Σήμερα έχουμε ένα οργανισμό συνοριοφυλακής ακτοφυλακής ολοκληρωμένο, ε, ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων, και συστήματα πληροφόρησης που γίνονται διαλειτουργικά όλο και περισσότερο. Με τον νέο κανονισμό που συζητούμε σήμερα θα μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Ένα στοιχείο κλειδί είναι το μόνιμο σώμα συνοριοφυλάκων ακτοφυλάκων που θα δημιουργηθεί γρήγορα και θα αναπτύξει την πλήρη επιχειρησιακή ε, δυνατότητα των 10.000 ατόμων μέχρι το 2027. Όμως θα μπορούμε να παρακολουθούμε ήδη την 1η Ιανουαρίου του 2021 ε, την ε, αύξηση του προσωπικού. Το άλλο στοιχείο κλειδί που αλλάζει τα πράγματα είναι ότι το μόνιμο προσωπικό του οργανισμού θα έχει εκτελεστικές εξουσίες. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορεί να κάνει διαχείριση συνόρων, καθήκοντα επιστροφών, αυτοδικαίως. Βέβαια, οι αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής θα παραμείνουν υπεύθυνες και θα διοικούν και θα ε, είναι επικεφαλής στις δραστηριότητες των οριοφυλάκων και ακτοφυλάκων που λαμβάνουν χώρα στο έδαφος τους ενώ θα είναι ε, υπό το κράτος μέλος υποδοχής, κάποια ε, ε, θα υπάρχει δυνατότητα να γίνεται έλεγχος σε έγγραφα ταυτοτήτων, να υπάρχει άρνηση της εισόδου, να σφραγίζονται τα ταξιδιωτικά έγγραφα, να σταματούνται άτομα που παράτυπα επιχειρούν να περάσουν τα σύνορα και να υπάρχει και ε, υποστήριξη σε διαδικασίες επιστροφών και από άλλες ε, χώρες, από προσωπικό από άλλες χώρες ε, ή για υπηκόους που επιστρέφουν με αναγκαστικά μέτρα. Θα πρέπει επίσης να διασφαλιστεί ότι θα εφαρμόζονται και θα γίνονται σεβαστά τα ε, υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και θα υπάρχει σωστή ε, κουλτούρα επιχειρήσεων. Ο οργανισμός θα στηρίζει περισσότερο τα κράτη-μέλη στις επιστροφές για να βελτιώνεται η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ε, εμένουσες προκλήσεις μεταναστευτικές. Χαιρετίζω κι άλλες εξελίξεις που συμφωνήθηκαν στα πλαίσια αυτού του κανονισμού όπως εξυγχρονισμός του παρακολούθηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στα πλαίσια της επιχειρησιακής δραστηριότητας του οργανισμού. Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι στην καρδιά όλων των πρωτοβουλειών της Κομισιόν και αυτής. Όλες οι δραστηριότητες του οργανισμού και των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών θα σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα τα οποία θεσπίζονται στο χάρτη. Ο οργανισμός θα συνεργαστεί στενά με τον μελλοντικό οργανισμό ασύλου για να έχει πρόσβαση στις διαδικασίες του ασύλου. Ο οργανισμός θα βοηθήσει να διασφαλίσουμε επίσης ότι εκείνοι που δεν χρήζουν διεθνούς προστασίας θα επιστρέφονται με πλήρη σεβασμό τον, επαναλαμβάνω αυτό, ε, πλήρη σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Ελπίζω ότι όταν θα συγκροτηθεί το επόμενο κοινοβούλιο, η πρόταση σύστασης ε, του, οργανισμού, ε, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασύλου θα εγκριθεί σύντομα. Ελπίζω. Θέλω επίσης να προσθέσω ότι λυπάμαι διότι η δυνατότητα μηνιαίας διαφορικής πληρωμής στο μόνιμο προσωπικό η πρόταση αυτή δεν διατηρήθηκε στην τελική συμφωνία. Αυτό είχε στόχο να βελτιώσει την ελκυστικότητα του οργανισμού ως εργοδότη, να διασφαλίσει επίσης μόνιμο προσωπικό που θα προσλαμβάνεται έγκαιρα. Ε, σχετικά με αυτό θα δώσω μια διακήρυξη. Τέλος, πολιτική καθοδήγηση για την ε, ε, ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων. Αυτό σημαίνει σχεδιασμό ικανοτήτων για τον οργανισμό συνοριοφυλακής και ακτοφυλακής, ε, αυξημένη ε, συνέπεια με τις υπόλοιπες εξωτερικές πολιτικές της Ένωσης. Με αυτό τον καινούριο κανονισμό και ο οργανισμός και τα κράτη-μέλη θα έχουν εργαλεία για να αντιδρούν και να προβλέπουν μελλοντικές κρίσεις στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Τέλος, θα βοηθήσει αυτό στη διατήρηση της, ε, ε, του χώρου Σέγγεν ελεύθερης διακίνησης. Θα βοηθήσει στη διατήρηση του χώρου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Γκάιερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αξιότιμη επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Αναμφίβολα η νέα εντολή για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλάκων Ακτοφυλάκων είναι σημαντικό βήμα ε, ως ευρωπαϊκή αντίδραση για το μεταναστευτικό. Ε, προβλέπεται αύξηση σε 10.000 άτομα, ε, ε, πλοία, αεροσκάφη. Ε, έτσι θα μπορέσει να είναι πιο λειτουργικός οργανισμός και να σώζει και ζωές. Χρειάζονται πόροι. Γι' αυτό αυτό θα λειτουργήσει μόνο αν ε, συμφωνήσουμε σε ένα δημοσιονομικό πλαίσιο πολιετές και διευρυμένο. Και εδώ θα ήθελα να αναφερθώ στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Αυστρίας, για παράδειγμα, θα ήθελα να πω ότι όποιος θεωρεί σημαντική τη φύλαξη των συνόρων θα πρέπει να πληρώσει και ε, μεγαλύτερο προϋπολογισμό. Αυτό είναι κομμάτι μόνο μιας συνεκτικής ευρωπαϊκής πολιτικής για την μετανάστευση και σίγουρα είναι και ε, μια πολιτική που εκφράζει ε, αλληλεγγύη επίσης ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των προσφύγων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κοέλιο, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε και Επίτροπε, κύριε Βραμόπουλε, αγαπητοί συνάδελφοι. Η έγκριση αυτή τη νέα ενισχυμένη ενεργοφυλακή ακτοφυλακή είναι ένα ιστορικό βήμα για μια κοινή προστασία των εξωτερικών μα συνόρων. Σχετίζεται με την ελεύθερη κυκλοφορία ε, στον χώρο Σέγγεν. Μιλάμε για 10.000 ακτοφυλακέ που μπορούν να μεταφερθούν ε, στις χώρες όπου είναι πιο ευάλωτα τα σύνορα ή όταν προκύπτει κάτι επίγον. Αυτό δεν πρέπει βεβαίω να οδηγεί στα κράτη-μέλη να μην τηρούν τις ε, ε υποχρεώσεις τους. Τα, μισά από τα άτομα αυτά, από του οκτωφύλακε, θα προέρχονται από τα κράτη-μέλη. Η Πορτογαλία θα είναι έτοιμη το 2021 να στείλει 110 ε, συνοριοφύλακες. Ε, όμως, παραδείγματος χάρη, κάνουμε κάτι, κάποιες υποσχέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις οποίες ενδεχομένως τα κράτη-μέλη δεν μπορέσουν να τηρήσουν στη συνέχεια. Οι... Θα έχουν επίσης έναν ισχυμένο ρόλο ε, για την επιστροφή ανθρώπων που παραμένουν παράνομα στη χώρα μας. Το ένα τρίτο των αποφάσεων όμως εφαρμόζονται, των αποφάσεων, αποφάσεων επιστροφής. Για την Πορτογαλία δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία. Επίσης ε, υπάρχει το θέμα των δευτερογενών μεταφορών μεταφορών, μετα, μετα ε, βιβάσεων και έχουμε δει ότι τέσσερα κράτη-μέλη χωρίς κανένα απολύτως λόγο κατάργησαν τη Σέγγεν. Ε, και να πω κάτι τελευταίο έκανε για τον εισηγητή που κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ πολύ για δύο λεπτά ο κύριος Νίντερ Μιούλερ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια, τη Ρομπέρτα Μέτσολα, για την πολύ επικοδομητική συνεργασία που είχαμε, χωρί την οποία δεν θα είχαμε καταφέρει να εκπονήσουμε αυτή την νομοθετική πρόταση. Να ευχαριστήσω όμω και τον Επίτροπο, τον κύριο Αβραμόπουλο, και όλο το προσωπικό του γραφείου του για την πολύ στεναρή υποστήριξή του το 2015 αυξήθηκε δραματικά ο αριθμό των μεταναστών που φτάναν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν επιτακτική λοιπόν η ανάγκη να ενισχύσουμε την προστασία των εξωτερικών συνόρων. Κατά συνέπεια, το 2016 είχαμε τη νέα πρόταση για τον Frontex. Η υφιστάμενη πρόταση αποτελεί μια θεωρωμένη πρόταση τη προηγούμενη πρόταση Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπω ακούσαμε, αυξάνεται το πεδίο εφαρμογή του οργανισμού πλέον και δίδονται περισσότεροι χρηματοδοτικοί πόροι, καθώ επίση και περισσότεροι εμπειρογνώμονε και μεγαλύτερο προσωπικό. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, πιστεύω, κατά τη διάρκεια των πραγματεύσεων να διασφαλίσουμε ότι ο Frontex θα εξακολουθήσει να σώζει ζωές όσων διακινδυνεύουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να υπολοιπόμεθα από την βασική μας αυτή ανθρωπιστική υποχρέωση. Δεν μπορεί ποτέ κυβερνήσεις, υπουργοί να παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές για εσωτερικού καθαρά πολιτικούς λόγους. Παράλληλα τώρα η πρόταση αυτή δίνει στον οργανισμό αυτό περισσότερες αρμοδιότητες στην εφαρμογή των επιστροφών, για όσους δηλαδή δεν έχουν καταφέρει να πάρουν άσυλο. Αυτό όμως θα πρέπει να ισχύει μόνο για τους πρόσφυγες στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θα πρέπει να δίδεται καμία νομική δυνατότητα στον οργανισμό να συμμετέχει σε επιστροφές από μία τρίτη χώρα προς μία τέταρτη χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να διασφαλίσουμε ότι η πρόταση αυτή θα ενισχύει τι υποχρεώσει και τι δεσμεύσει του οργανισμού αυτού όσον αφορά τα ανθρώπινα και θεμελιώδη δικαιώματα. Τέλο, είναι λυπηρό το ότι ε, ενώ καταβάλαμε προσπάθειε για να προστατεύσουμε καλύτερα τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, το Συμβούλιο από την άλλη δεν κατάφερε να καταλήξει μια συμφωνία όσον αφορά το κοινό σύστημα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μεταρρύθμιση του συστήματο του Δουβλίνου παρεμποδίστηκε τελικά λόγω καθαρά εσωτερικών πολιτικών λόγων και νομίζω ότι ε, και η έγκριση της προκαταρκτικής συμφωνίας ε, όσον αφορά την υπηρεσία αυτή τελικά δεν ευωδόθηκε λόγω εσωτερικών εθνικών εγωισμών. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε, και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και από την έκθεση, ένα ευρωπαϊκό ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των συνόρων και αυτό σαφώς θα απασχολήσει και την επόμενη νομοθετική θητεία. Ο κύριος Βίστησεν τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Τα εξωτερικά σύνορα ε, έως τώρα από ό,τι φαίνεται ποτέ δεν ήταν αντικείμενο ε, πραγματικής ε, προστασίας. Αυτό μας λέτε σήμερα με αυτό το νομοθέτημα. Γι' αυτό το λόγο 18 χρόνια μετά τη Σέγγεν ήρθε η ώρα νομίζω να έχουμε μια υπηρεσία συνόρων. Ο λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε το συμβασμό που προέκυψε τον Τρίλογο είναι ότι φοβούμαστε ότι είναι πολύ λίγα αυτά που προτείνεται και έρχονται πολύ αργά. Πολλές δικλείδες ασφαλείας ε, δεν θα έχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα για την ασφάλεια των Ευρωπαίων. Δεν μπορείτε να βοηθήσετε την επιστροφή σε τρίτες χώρες. Ε, αυτή τη στιγμή εγκρίνουμε μία λύση η οποία όμως δεν θα ικανοποιήσει κανέναν, ούτε τους πολίτες, ούτε θα είναι πιο ασφαλέ το Σέγγεν. Ευχαριστώ κυρία Γκρίσπα για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Το Σεπτέμβριο του 2018 ο πρόεδρος Γιούνκερ παρουσίασε μια νέα μεταρρύθμιση της υπηρεσία Frontex. Και πριν από δύο χρόνια ε, ήμουν εισηγήτρια και είχα χαιρετήσει ε, την το αποτέλεσμα τη πρώτη αναθεώρηση. Στο όνομα τη ομάδα μου σήμερα κάνω πάλι το ίδιο. Σε ένα πολύ μικροχρονικό διάστημα, σε ένα χρόνο ρεκόρ. Λυπάμαι βέβαια ε, για κάποια σημεία. Παρ' όλα αυτά είμαι ικανοποιημένη για το πόσο γρήγορα μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε την εξέταση του ζητήματο αυτού με μια ισορροπημένη προσέγγιση, αποτελεσματική για την προστασία των συνόρων μα, σεβόμενη τα θεμελιώδη δικαιώματα ε, όπω μα το ζητούσαν οι συμπολίτε μα σημειώνω κυρίω και χαίρομαι γι' αυτό ότι γίνεται ένα πραγματικό βήμα προ τα μπρο σε δημοσιονομικό επίπεδο, σε επίπεδο δυνατοτήτων δηλαδή, αλλά και σε επίπεδο αρμοδιοτήτων, όπω μόλι αναφέρθηκε. Δύο στοιχεία θα ήθελα όμω να τονίσω. Χαίρομαι που λαμβάνουμε γνώση τη δημιουργία μια μόνιμη δύναμη που θα αποτελείται από 10.000 ακτοφύλακε και συνοριοφύλακε και όπου τα κράτη-μέλη θα οφείλουν να συνεισφέρουν είναι πιο αξιόπιστο, πιο αποτελεσματικό, πιο συγκεκριμένο από αυτήν, το, αυτό το απόθεμα των 1500 ανθρώπων που είναι διαθέσιμο υποτίθεται, αλλά με ένα σύστημα που δεν λειτουργεί. Είναι λοιπόν ένα χρήσιμο, ένα απαραίτητο βήμα και συγκεκριμένο. Δεύτερον, ε, ω εισηγήτρια στην αναθεώρηση, είχα ζητήσει στο τελικό κείμενο να γίνει μια αναφορά στη δημιουργία ενό κέντρου κατάρτιση Frontex. Διότι αν θέλουμε να ξεπεράσουμε ε, την εθνική ε, προσέγγιση για την προστασία των συνόρων, διότι τα κράτη-μέλη προφανώ και είναι αρμόδια και παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Όμω, εάν θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί στον ευρωπαϊκό χώρο ελεύθερη κυκλοφορία, τη Σέγγεν δηλαδή, εάν θέλουμε να είναι όσο γίνεται λιγότερα τα κενά, πρέπει να είμαστε Ευρωπαίοι. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα εργαλείο ευρωπαϊκό. Και η υπηρεσία θα πρέπει να μπορεί να συνεργαστεί με τις αρχές των κρατών μελών. Όχι μόνο να, τι υποστηρίζει, να συνεργάζεται μαζί τους. Για να μπορεί να γίνει όμως αυτό στην πράξη θα πρέπει να αναπτύξουμε μια, μια πραγματική ευρωπαϊκή κουλτούρα σε επίπεδο κατάρτισης. Αυτό ακριβώς ε, ζητεί το κείμενο και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τη Ρομπέρτα Μετσόλα, την εισηγήτρια, η οποία έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, έδειξε μεγάλη ενέργεια, αποφασιστικότητα και χάρη σε αυτήν μπορούσαμε να προχωρήσουμε γρήγορα. Σε λίγες ώρες ε, η ομάδα μου θα υποστηρίξει στην ψηφοφορία αυτήν τη νέα μεταρρύθμιση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Αλμπιόλ Γκούθμαν. Έχει το λόγο για ένα λεπτό. Τελειώνει αυτή η θητεία και, και ουσιαστικά όσοι κυβερνούν την Ευρώπη έχουν εγκαταλείψει οποιαδήποτε ανθρωπιά. Πολιτικές που βασίζονται ουσιαστικά στον θάνατο των ανθρώπων στη θάλασσα, ε, στη σκλαβιά τους, ε, τις, ε, τα βασανιστήρια σε κέντρα κράτηση και τον εκτοπισμό του σε χώρε όπου δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα γίνουν σε αυτά τα δικαιώματά του. Είναι σκληρό αυτό που λέω, αλλά είναι αλήθεια. Αυτή είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπάρχουν ε, ε, τρόποι εισόδου νόμιμοι και ασφαλεί. Δεν υπάρχουν ανθρωπιστικέ θεωρήσει. Πλέον δεν επιτρέπουμε καν στι μη κυβερνητικέ οργανώσει να κάνουν τη δουλειά αυτή, η οποία είναι απαραίτητη. Κάποια στιγμή θα, θα περάσουν από δίκη οι πολιτικοί δίνονται για τις πάνω από 17.000 νεκρούς των τελευταίων 5 ετών στη Μεσόγειο. Οι πολιτικές τους που κλείνουν τα σύνορα και που ε, ουσιαστικά υποχρεώνουν τους μετανάστες να παίξουν τη ζωή τους γράμματα οδηγούν στο θάνατο 10 ατόμων τη μέρα. Και ο κανονισμός που ε, ψηφίστε σήμερα ουσιαστικά είναι το απάβγασμα αυτής της απάνθρωπης πολιτικής. Είναι ένα ε, μια παραστρατιωτική οργάνωση με 10.000 ανθρώπους με 2 δισεκατομμύρια ευρώ προπολογισμό για να ε, κλειδαπαρώσουν τα σύνορα, για να εκτοπίσουν τους ανθρώπους, για να κλείσουν τους ανθρώπους σε κέντρα ε, ε κράτησης. Είναι ουσιαστικά το ο στρατιωτικός βραχίωνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το όνειρο της ακροδεξιάς που το κάνουν πραγματικότητα φιλελεύθεροι σοσιαλιστές και συντηρητικοί. Η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την καλή συνεργασία και την ολοκληρωμένη προσέγγιση. Νομίζω ότι είχαμε πολύ επικοδομητική θέση ως Κοινοβούλιο, ιδιαίτερα στη διάσωση και την έρευνα. Εμείς ε, φροντίσαμε η Frontex να έχει κατάλληλη εντολή έρευνας διάσωσης λόγω της ανθρωπιστικής κρίσης που βλέπουμε να ε, ε, λαμβάνει χώρα στη Μεσόγειο. Η πλειοψηφία ετάχθη πέρα αυτών. Αλλά τα κράτη-μέλη ψήφισαν διαφορετικά. Ε, μπλοκάρισαν τις προσπάθειες της εισηγήτριας να ενισχύσουν τη διάσωση στο κείμενο του νομοθετήματος. Και αυτό είναι πρόβλημα πραγματικό. Η Frontex μπορεί να διασώζει μόνο ανθρώπους στα πλαίσια και στα, μέσα στα όρια της επιχείρησης διάσωσης και ε, είναι πολύ μικρή περιοχή, λίγο έξω από τη Σικελία. Δεν είναι αυτή η περιοχή όπου υπάρχει το πρόβλημα. Και πνίγεται κόσμο στη Μεσόγειο τώρα που μιλάμε και παρακολουθούμε. Ξέρουμε που είναι. Συ... Οι δεδαγμένες είναι σαφείς. Κανείς δεν πάει όμως να διασώσει αυτούς τους ανθρώπους. Ε, οι κυβερνητικές οργανώσεις ε, ε, ποινικοποιούνται, τους παίρνουν τα πλοία, δεν γίνονται επιχειρήσεις και η ε, ε, έρευνα και διάσωση ε, έγινε στη, κοντά στη Λιβύη, αλλά διασώσεις δεν γίνονται, γιατί τώρα ξέσπασε πόλεμος πάλι εκεί. Έτσι παραβιάζεται η υποχρέωση διάσωσης ε, μακροπρόθεσμα πρέπει να υπάρχει στη Μεσόγειο ε, οργάνωση σε επίπεδο κρατών μελών. Ε, ε, τα κράτη-μέλη δεν, να, δεν είναι διατεθειμένα να βοηθήσουν. Θα πρέπει λοιπόν να εργαστούμε με συντονισμένο τρόπο, αλλιώς θα καταρρεύσουν οι αξίες της Ευρώπης μαζί με τους πνιγμένους. Δέχεστε μπλε κάρτα κυρία Κέλλερ. Όχι. Λυπάμαι, προσπάθησα πάντως. Η κυρία Τζέιμις τώρα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Mike, Mike. Μικρόφωνο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μάταιες προσπάθειες να αντιμετωπίσει μια πολιτική μετανάστευση ε, χωρίς νόημα. 11 ε, δις ευρώ δαπανώνται ε, γι' αυτό. Ο Φραντ Τίμερμανς είπε τον περασμένο μήνα ότι η Ευρώπη δεν